12 ε, εκ νέου αρχίσασα. Τα πρακτικά της συνεδρίας 20 Απριλίου 2012 έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις. Εάν όχι, θεωρούνται τα πρακτικά ότι έχουν εγκριθεί.